υπόλοιπες ερωτήσεις. Λίγη ο χρόνος για ε, συνεδρίαση και η επόμενη συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 9 ε, μέχρι τη 1 και 3 ε, με 7. Υπάρχει η, η μέρη διάταξη που έχει δημοσιευθεί